More generally, reforms have however continued agenda. Οι μεταρρυθμίσεις όμως συνεχίστηκαν και το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει στρατηγική προτεραιότητα της χώρας. Ο διάλογος υψηλού επίπεδου για την ένταξη είναι χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα συνεχίσει να εστιάζει σε βασικά θέματα συμπεριλαμβανομένων των καλών σχέσεων, των σχέσεων καλής γειτονίας. Αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαπραγματεύσεις ένταξης. Η προτεραιότητα για τον επόμενο χρόνο θα πρέπει να είναι η αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή των υπαρχών των νομικών και πολιτικών πλαισίων. Ε, σημαντική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο κράτος δικαίου και στην επίτευξη αποτελεσμάτων από την πάλη κατά των οργανωμένου εγκλήματος. Η ελευθερία έκφρασης επίσης παραμένει ένα θέμα που απασχολεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει την έναρξη διαπραγματεύσεων ένταξης για πέμπτη φορά δεν έχει ληφθεί απόφαση μέχρι σήμερα από το Συμβούλιο. Ε, μία ανάληψη δράσης ε, συνεπάγεται τον κίνδυνο να υπονομευθούν και οι μεταρρυθμίσεις στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και να υπονομευθεί και η ε, αξιοπιστία της πολιτικής διεύρυνσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη, όπως ήταν πάντοτε, να παρουσιάσει πρόταση για διαπραγματευτικό πλαίσιο χωρίς, χωρίς ε, αναβολή, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να ληφθεί το θέμα του ονόματος σε πρώιμο στάδιο στις διαπραγματεύσεις ένταξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αν η οι πρώτες ε, συζητήσεις, ε, η πρώτη εξέταση και οι συζητήσεις του Συμβουλίου για το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ε, είχαν αρχίσει, θα είχε δημιουργηθεί η απαραίτητη δυναμική η οποία θα υποστήριζε την εξέβρεση λύσης για το όνομα ακόμα και πριν ανοίξουν τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων η εφαρμογή της νέας προσέγγισης στα κεφάλαια 23 και 24 θα έδινε τα ε, μέσα, τα εργαλεία, ούτως ώστε να καταπιαστούμε με βασικά θέματα που απασχολούν τα κράτη-μέλη. Στην Αλβανία υπήρξε σημαντική πρόοδος ε, την περίοδο μέχρι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου δύο βασικά νομοθετήματα και ο εσωτερικό κανονισμός του Κοινοβουλίου εγκρίθηκαν με διαπαραταξιακή υποστήριξη. Οι εκλογέ έγιναν ομαλά και ο λαός έδωσε σαφή εντολή στου ηγέτε του. Ε, δεδομένου ότι η Αλβανία ολοκλήρωσε την απαραίτητη πρόοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει ε, να χορηγήσει το Συμβούλιο στην Αλβανία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας με τη συμφωνία ότι η Αλβανία θα συνεχίσει να καταπολεμεί το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθαρά. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει την έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης, η Αλβανία θα πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες που ήδη έγιναν και να αναλάβει δράση, ούτω ώστε να ασχοληθεί ε, σε βάθος με τα εξής πέντε θέματα προτεραιότητες. Πρώτον, να συνεχίσει να εφαρμόζει την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Δεύτερον, να αναλάβει περαιτέρω δράση για να ε, πραγματοποιήσει την ανεξαρτησία, αποτελεσματικότητα και λογοδοσία ε, δικαστικής εξουσίας. τρία Να καταβάλει περαιτέρω αποφασιστικές προσπάθειες στην καταπολέμηση της διαφθοράς. τέταρτον Να καταβάλει περαιτέρω αποφασιστικές ε, προσπάθειες στην ε, μάχη για ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα και πέμπτον να αναλάβει αποτελεσματικά μέτρα για να ενισχύσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των Ρωμά και ε, πολιτικές κατά των διακρίσεων όπως και για την εφαρμογή των ε, ε, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει τις προσπάθειες της Αλβανίας προς την επίτευξη αυτών των προτεραιοτήτων των βασικών, ε, αρχίζοντας ένα διάλογο υψηλού επίπεδου με την χώρα. Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι σε στασιμότητα. Χθες το βράδυ η ποδοσφαιρική ομάδα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ε, έδειξαν έντονο ομαδικό πνεύμα και ενότητα και εξασφάλισαν μια νύχτα επιτυχίας, ε, μια νύχτα ε, επιτευγμάτων. Τώρα έχουμε στην Ευρωπαϊκή, μια Ευρωπαϊκή ομάδα στο Σαράγεβο που προσπαθεί να στηρίξει τα πολιτικά κόμματα, να στηρίξουν την ε, απόφαση για την υπόθεση Sage Dick που θα άνοιγε νέα εποχή για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και τους πολίτες της. Το μήνυμά μου σήμερα στους πολιτικούς της Βοσνίας είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των ποδοσφαιριστών σας, να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των πολιτών σας, να τους ε, παραδώσετε ένα νέο μέλλον. Εμείς έχουμε αναλάβει δέσμευση να βοηθήσουμε, αλλά η περαιτέρω πρόοδος εξαρτάται από την ικανότητα των πολιτικών ηγετών να συμφωνήσουν μαζί σε μια συμβιβαστική λύση που θα ανοίξει το δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα βοηθήσει να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα των ηγετών τους να ε, προωθήσουν την ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, προλιάνουν το έδαφος για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και μετά για μια αξιόπιστη, ε, ένα αξιόπιστο αίτημα ε, προσχώρησης. Το 2013 η απόφαση του Συμβουλίου που εξουσιοδοτεί την έναρξη ε, των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης έφερε το κοσυφοπαίδιο σε μια νέα σημαντική φάση στην Ευρω... στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοσυφοπεδίου. Αυτό αποτελεί αναγνώριση της προόδου που έγινε σε βασικές μεταρρυθμίσεις και στις σημαντικές, των σημαντικών προσπαθειών που έγιναν από το Κωσυφοπέδιο προς την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Σερβία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να ολοκληρωθεί τις διαπραγματεύσεις την Άνοιξη του 2014 και να μονογραφήσει τη συμφωνία σχέδιο το καλοκαίρι. Μετά θα υποβάλει τις προτάσεις ε, προς υπογραφή από το Συμβούλιο για να συναυθεί η συμφωνία και κύριε Πρόεδρε βεβαίως θα σας κρατώ ενήμερος σχετικά με την εξέλιξη ε, στις διαπραγματεύσεις για το Συμβούλιο σταθεροποίηση και σύνδεση σε όλα τα βασικά στάδια των συζητήσεων. Το Κωσυφοπαίδιο κατέλαβε προσπάθειε να διασφαλίσει την πρόοδο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων και αυτό το διατήρησε υψηλά στο πολιτικό του θεματολόγιο από την πλευρά μα. Επίσης ε, εμένουμε στη δέσμευσή μας και προτιθέμεθα να ε, υποβάλλουμε έκθεση για στο πρώτο εξάμεινο του 2014 για την πρόοδο. Τώρα το Κωσυφοπαίδιο θα πρέπει να στηρίξει ενεργά την Γιούλεξ για να εφαρμόσει την εντολή της. Επίσης θα πρέπει να εστιάσει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ε, που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του ε, βάσει ενός μελλοντικού, μιας μελλοντικής συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. Πολύ σημαντικό είναι εδώ το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά. Επίσης, κονδύλια από το προενταξιακό μέσο θα βοηθήσουν στην υλοποίηση της συμφωνίας του Απριλίου που θα συμπεριλαμβάνουν και την υποστήριξη των σερβικών κοινοτήτων στο Κωσυφοπαίδιο. Η Τουρκία αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της οικονομίας της και το σημαντικού ρόλου που παίζει στην εξωτερική πολιτική και την ε, ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια. Ε, το θετικό θεματολόγιο ε, που άρχισε το 2012 συνεχίζει να στηρίζει και να συμπληρώνει τις διαπραγματεύσεις ένταξης. Ε, σημειώθηκε πρόοδος ε, στις ε, δικαστικές μεταρρυθμίσεις και η κυβέρνηση άρχισε μια ιστορική ειρηνευτική διαδικασία με στόχο τον τερματισμό της τρομοκρατίας και της βίας στην νοτιοανατολική Τουρκία, εξομαλύνοντας έτσι το δρόμο για λύση του κουρδικού ζητήματος. Οι διαδηλώσεις το Μάιο και τον Ιούνιο και η υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία ε, καθώς και η πλήρης απουσία διαλόγου δημιούργησαν σοβαρές ανησυχίες. Ε, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι έρευνες ε, σχετικά με τη συμπεριφορά της αστυνομίας και όσοι φέρουν ευθύνες να λογοδοτήσουν. Εγώ άκουσα τις φωνές που έλεγαν ότι η σωστή απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα επεισόδια στο Γκέζι Πάρκα θα πρέπει ε, να είναι ε, να απεμπλακεί η Ένωση. Αλλά το μήνυμα του πακέτου που εγκρίθηκε σήμερα είναι διαφορετικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τη δέσμευσή της και να συνεχίσει να στηρίζει την Τουρκία και τους Τούρκους πολίτες να ε, ολοκληρώσουν τις ε, θεμητές προσδοκίες τους ε, περαιτέρω μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την ελευθερία της έκφρασης των μέσων και την ελευθερία του συναθρίζεσθε η δέσμη εκδημοκρατισμού που παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2013 ε, συνεπάγεται μια προοπτική προόδου επί σειράς θεμάτων συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γλωσσών άλλων από της τουρκικής. Ε, επίσης λαμβάνονται υπόψη και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Όπως ανέφερα, ε, η πλήρης δυναμική των σχέσεών με στην Τουρκία θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο στα πλαίσια μιας διαδικασίας ενεργού ε, και αξιόπιστης προς την ένταξη όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει ε, το συγκριτικό σημείο αξιολόγησης για τις μεταρρυθμίσεις. Έχουμε πάρα πολλά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η ε, υπογραφή της ε, Συμφωνίας ε, Επανεισδοχής ε, Θεωρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και η έναρξη της, δια, της διαδικασίας απελευθέρωσης από των θεωρήσεων ταυτόχρονα θα είναι μια κατάσταση που θα επιφέρει ωφέλη και για τις δύο πλευρές και η Επίτροπος Μάλμστρομ και εγώ έχουμε αναλάβει πλήρη δέσμευση εδώ. Τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο της Τουρκίας. Ας παίξει μπάλα. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, ούτω ώστε ε, πολύ συγκεκριμένα να καταδείξουμε τα πλεονεκτήματα μια σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία στου Τούρκου πολίτε. Θέλω επίση να υπογραμμίσω τη σημασία τη προόδου στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκία και όλων των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένη τη Δημοκρατία τη Κύπρου. Τώρα είναι κατεπήγον η Τουρκία να ε, ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της της πλήρους εφαρμογής του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου. Ε, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει από την Ελληνοκυπριακή και την τουρκο κοινότητα να ε, ξαναρχίσουν ε, πλήρως τις διαπραγματεύσεις για μια συνολική λύση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς ε, ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να κάνουν ό,τι, είναι δυνατόν για να εδρεωθεί θετικό κλίμα μεταξύ των κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι έτοιμη να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την υποστήριξή της για τη διαδικασία αυτή, ε, αν το ζητήσουν τα δύο μέρη και αν συμφωνήσουν τα Ηνωμένα Έθνη. Με την απόφαση της νέας κυβέρνησης της Ισλανδίας να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη, η διαδικασία ένταξης ε, πέρασε σε περίοδο στασιμότητας. Όμως θα πρέπει να είμαι απόλυτα ε, ξεκάθαρος. Η Ισλανδία παραμένει σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις μας ανα πάσα στιγμή. Από τη δική μας την πλευρά δεν έχουμε απεμπλακεί. Οποτεδήποτε και αν κάποτε η Ισλανδία θελήσει να το κάνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις εργασίες επί των διαπραγματεύσεων που έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο. Και εξακολουθώ να ε, είμαι αισιόδοξο ότι θα φτάσουμε σε ένα υποφελές αποτέλεσμα θετικό για όλες τις πλευρές. Κύριε Πρόεδρε, ε, παρουσίασα μια εικόνα σήμερα μιας ε, ισχυρής και ανοιχτής διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολείται με τα θεμελιώδη πρώτα. Μια διαδικασία όπου οι υποψήφοι και οι δυνάμοι υποψήφοι θα οικοδομούν την αξιοπιστία τους μέσα από επιδόσεις στις μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμόζονται και θα υλοποιούνται. Ε, βλέποντας ε, το έργο που μας περιμένει του χρόνου, ε, θεωρώ ότι η συνεργασία και η υποστήριξη αυτής της Επιτροπής θα απαιτηθεί περισσότερο από ποτέ, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα ωφέλη και οι ευκαιρίες από τη διεύρυνση θα συνεχίσουν σταδιακά να οικοδομούνται μέχρι την ένταξη και πέραν αυτής. Προσβλέπω στην ε, αντίδραση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάθε, σε κάθε μία από τις ε, εκθέσεις των χωρών και περιμένω τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Δύο λεπτά θα έχουν οι συγητέ και οι άλλα δύο οι συγητές. Μην ξεπεράσετε το χρόνο για να δοθεί χρόνος και σε άλλους συναδέλφους, ιδιαίτερα στους τρεις συναδέλφους που κούκαν φλότρε και Ρουζέκα που είναι επικεφαλής ε, αντιπροσωπιών που θα έπρεπε να, ε, πολιτικών ομάδων. Ε, Στην ε, Βοσνία Ερζεγοβίνη όμως πώς θα επιτελεστεί η πρόοδος ε, αν οι, ε, ο και ο ε, έχουν σουηδικά διαβατήρια. Στην περίπτωση της Αλβανίας δε έμαθα ότι με μία υπεύθυνη αντιπολίτευση μπορεί να κάνει πραγματικά μεγάλη διαφορά και αυτό το εννοώ με κάθε σοβαρότητα. Τώρα η κυρία Γκόμες, ο κύριος Αλαφράγκα, μετά από το ΕΛΚ. Κυρία Γκόμες. Δεν είναι εδώ. Εδώ είμαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σε σχέση με την Τουρκία, από ό,τι κατανοώ, από αυτά που είπατε, και με βάση το πακέτο μεταρρυθμίσεων που έχει επιτευχθεί κινείται προς την σωστή κατεύθυνση αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των Τούρκων δηλαδή των πολιτών που διαμαρτυρήθηκαν στο πάρκο Γκεζή. Πώς αντιλαμβάνεστε το θέμα και εκτιμώ αυτά που είπατε για την Κύπρο. Τι μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε τα συμβαλόμενα μέρη να συνδράμουν σε αυτές τις πλήρεις διαπραγματεύσεις για την Κύπρο. Ως προς το Κωσυφοπαίδιο, ε, πιστεύω ότι θα ανοίξει η συμφωνία πέντε μέρες πριν από τις εκλογές στο Κωσυφοπαίδιο. Τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει αυτό Δηλαδή φαίνεται ότι υποστηρίζουμε την ε, κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή κατέχει την εξουσία. Υπάρχει ίση εκπροσώπηση και δίκαιοι κανόνες παιχνιδιού. Μιλήσατε επίσης για τις ε, διμερείς ε, αντιγνωμίες που υπάρχουν και διαφωνίες τι επιπτώσεις θα υπήρχαν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των χωρών, ιδιαίτερα ως προς την ονομασία της ΦΥΡΟΜ. Πέντε κράτη-μέλη δεν έχουν αναγνωρίσει το Πέδιο. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε αυτή την... Ε, και ένα άλλο ζήτημα μιλήσατε για την μεταρρύθμιση στον τομέα, στο δικαστικό τομέα και την καταπολέμηση του εργονομένου εγκλήματος. Πώς μπορούμε να δράσουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον ατιμορρησία αυτών που εμπλέκονται ε, σε σχέδια διαφθοράς. Διότι αυτό το βλέπουμε και εντός ευρωπαϊκού εσωτερικού χώρου. Ο κύριος Κούκαν από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Φίλε, διότι μας παρουσίασε το πακέτο και την έκθεση πρόοδου. Και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι γιατί έχει πραγματικά εντρυφήσει σε αυτό το θέμα της ε, ενταξιακής διαδικασίας και ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Από ό,τι είπατε κύριε Επίτροπε, καθίσταται σαφές ότι η διαδικασία διεύρυνσης προωθείται στα Δυτικά Βαλκάνια. Η κατάσταση είναι διαφορετική σε κάθε χώρα. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά νέα. προσπαθούμε με κάθε μέσο να βρούμε κάτι θετικό να πούμε για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το μόνο θετικό ήταν το αποτέλεσμα του ποδοσφαίρου. Τώρα για να μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά. Αυτή η διαδικασία δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει σοβαρό ρόλο στην περιοχή και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επηρεάσει αυτές τις χώρες στην αναπτυξιακή τους πορεία. Θα πρέπει να αυξήσουμε και την αξιοπιστία μας στην περιφέρεια αυτή, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε αξιόπιστους εταίρους σε συγκεκριμένες χώρες. Υπάρχουν παραδείγματα όπως ο διάλογος Σερβίας-Κωσυφοπεδίου, που θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Κύριε Επίτροπε, στην ομιλία σας μιλήσατε για τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Δεν είναι αυτό τυχαίο στην όλη διαδικασία. Πολλές φορές πρέπει να γυρίσουμε στο πρώτο τετραγωνίδιο. Επίσης μιλήσατε για εφαρμογή. Βεβαίως θα πρέπει να το προωθήσουμε και όχι οποιαδήποτε τύπο ε, εφαρμογή implementation. Με αγριοκοιτάει ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να ε, φέρω, σε, φέρω σε δύσκολη θέση, γι' αυτό θα σταματήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η πρώτη συζήτηση. Θα έχουμε αρκετό χρόνο για να μπούμε σε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Η κυρία Νέιτς από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εξ ονόματος της, Επιτροπή, της ομάδας μου και της αντιπροσωπείας μου σας ευχαριστώ πολύ για την συνολική εικόνα που μας παρουσιάσετε για την τρέχουσα διαδικασία διεύρυνσης. Έχετε δίκιο τονίζοντας ότι η διαδικασία διεύρυνσης βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια όπως τα κριτήρια της Κοπενχάγης σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, όμως έχει υποστεί μία, ε, ένα μετασχηματισμό. Ακούμε από υποψήφιες χώρες μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων ότι τα κριτήρια σήμερα είναι πιο αυστηρά από ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια. Αυτό ισχύει αλλά και η Ένωση δεν είναι η ίδια. Γι' αυτό θα πρέπει να προσαρμοστούμε στην, ε, στις αλλαγές αυτές. Έχετε μεγάλα χαρίσματα διπλωματίας, κύριε Επίτροπε, αλλά μιλήσατε για το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη και οι κυβερνήσει έχουν μείνει πίσω. Ενώ η Επιτροπή συνεχίζει προωθώντας τις προσφορήσεις αυτές και μας πείσατε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος έτσι ώστε οι χώρες αυτές να υποστούν αυτούς τους ε, μετασχηματισμούς και τις αλλαγές για να ε, βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών. Όμως οι κυβερνήσεις έχουν μείνει πίσω, γιατί είπαμε ότι πρέπει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Μακεδονία. Αυτό πρόθεσε η Κομισιόν, το έχει πει πέντε φορές, αλλά δεν έχει προωθηθεί. Εσείς είπατε ότι η Επιτροπή θέλει να δώσει ε, καθεστώς υποψηφιότητας και στην Αλβανία. Τέλος, εγώ αλλά και οι συνάδελφοί μου, κύριε Επίτροπε, συμφωνούμε μαζί σας ότι έχετε ασχοληθεί επικοδομητικά αλλά και ήσασταν επικριτικός εκεί που έπρεπε με τους εταίρους μας και αυτό είναι ύψης της σημασίας. Σας ευχαριστώ. Thank I'm standing for Εκπροσωπώ την κυρία Λούνατσεκ, η οποία δεν ε, βρίσκεται εδώ. Είναι σε μία αποστολή εκτός Βελγίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Μας παρουσιάσατε σαφέστατα και με αμεσότητα την κατάσταση ως έχει. Οι πράσινοι υποστηρίζουν τις συστάσεις της Επιτροπής. Επίσης θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριος Κούκαν για την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Έπρεπε να χρησιμοποιούμε ε, το καρότο και όχι το μαστίγιο σε αυτή τη ε, διαδικασία. Αλλά εάν ε, δεν λειτουργεί αυτή η προτρεπτική πολιτική, τότε δεν έχουμε και πολλές επιλογές, παρόλο που λυπάμαι ιδιαίτερα για τους πολίτες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ελπίζω το Συμβούλιο για μία φορά να ακούσει τις ε, συστάσεις της Επιτροπής και για την ΦΥΡΟΜ, καθώς και την Τουρκία. Ως προς το κοσυφοπέδιο, όπως είπε και, επειδή η κυρία Λούνατσεκ μάλλον είναι η συγγήτρια, ε, μας απασχολεί το θέμα της εκπνοής της εντολής του χρόνου. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα το αντιμετωπίσετε, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Εάν αποτύχουν οι εκλογές στο Βόρειο Κωσυφοπέδιο, τι θα γίνει. Επίσης, η εφαρμογή της συμφωνίας πώς θα εποπτευθεί μέσα στα πλαίσια του ανοίγματο των διαπραγματεύσεων. Γιατί δεν μπόρεσα να βρω το σωστό δρόμο μέσα από τα έγγραφα που έχω στη διάθεσή μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε και Επίτροπε, λάβαμε και την εισήγησή σας και χαίρομαι γι' αυτό. Έχω μία ανησυχία και ένα ερώτημα με απασχολεί το θέμα της Αλβανίας. Είμαι η Ιταλίδα. Πώς ξέρετε έχουμε πολλούς Αλβανούς ε, στην ε, παραοικονομία μας, ε, προβαίνουν σε εγκληματικές δραστηριότητες και επιδίδονται στην πορνεία και αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα στην Ιταλία. Είναι, αυτή είναι μία πτυχή, μία άλλη πτυχή των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν 50 εκατομμύρια άνθρωποι που θέλουν επίσης να εγκαταλείψουν την Αφρική γιατί δεν μιλάμε μόνο για εμπόλεμες σειράξεις αλλά δεν έχουν φαγητό αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν τρόφιμα. Τι θα κάνετε ως προς αυτή την πτυχή του θέματος, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που θα μεταβούν στην Ευρώπη. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ιταλικό και ευρωπαϊκό, έχει και μια παγκόσμια διάσταση, μια ευρύτερη διάσταση. Δεν είναι αστείο το θέμα, καθόλου αστείο. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ και εγώ τον Επίτροπο Διεύρυνσης και την ε, ολόκληρο το γραφείο του για τη δουλειά που έχω κάνει που είναι φανερώνεται πάρα πολύ μεγάλη. Ε, θέλω να πω ότι δεν έγινε μεγάλη αναφορά ε, στα θέματα της οικονομίας ε, των κρατών που είναι υποψήφια για ένταξη. Γιατί η οικονομία είναι η βάση της ευημερίας των, ανθρώπων. Και χωρίς να αμπαίνουμε στην ανάλυση της οικονομίας αυτών των κρατών και πώς θα αναπτυχθεί, ε, αλλά και για το γιατί να θέλουν να μπουν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με 25 εκατομμύρια φτωχούς και τόσους πολλούς άλλους κάτω από το όριο της στόχιας, Θέλω να πω με αυτό, πρέπει να εξετάσουμε το γεγονό ότι έχει πέσει το ενδιαφέρον των πολιτών και στην Ευρώπη αλλά και στα υποψήφια κράτη για ένταξη και αν είναι ακόμα στη διαδικασία της ένταξης δεν είναι γιατί θέλουν να μπουν, είναι γιατί φοβούνται να μείνουν απ' έξω. Πρέπει να μας απασχολήσει ε, το θέμα και της ηγεσία, όπως είπατε πριν για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αλλά νομίζω ότι έχει και ένα έλλειμμα ηγεσία γενικά η Ευρώπη. Ε, για την ε, Τουρκία είναι μια επανάληψη του ίδιου μοτίβου τα τελευταία δέκα χρόνια όπου καλείται η χώρα να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας το πρωτόκολλο. υπάρχει κανένα τρόπος να υποχρεωθεί ένα κράτος που δεν εφαρμόζει για δέκα χρόνια αυτό που την καλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει και είναι υποψήφια έτσι ώστε να εφαρμοστεί και η τελευταία μου ερώτηση. Η σημερινή Κυπριακή κυβέρνηση έχει πει πολλές φορές ότι ενδιαφέρεται να υπάρχει ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες για το Κυπριακό. Αναφερθήκατε στο Κυπριακό, είπατε για την εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών, δεν κάνατε καμία αναφορά για την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ερώτημα είναι, θέλετε, μπορείτε να σκεφτείτε έναν αντιπρόσωπο όπως το ζητάει η Κυπριακή Κυβέρνηση. Ναι. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για την παρουσίαση την οποία μας έκανε. Βεβαίω προσωπικά θεωρώ όταν η κυριαρχούσα τάση παγκοσμίω είναι η παγκοσμιοποίηση δεν μπορούμε να είμαστε κατά της διευρύνσεως. Πρέπει όμως η διεύρυνση να γίνεται με σωστό τρόπο σε τρόπο ώστε οι περιοχές, τα κράτη ε, που, που είναι υποψήφια προς ένταξη και προέρχονται από μια ειδική περιοχή και από πρώην ε, ένα ειδικό καθεστώς, κομμουνιστικό καθεστώς, πώς θα ενταχθούν με τον καλύτερο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα μπορέσουν να αφομοιωθούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποτελέσουν ε, ισότιμους εταίρους. Ε, από την έκθεση που μας είπατε και μας αναπτύξατε και από ε, την πρώτη ανάγνωση την οποία έκανα, πολύ πρόχειρη, βλέπω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε όλες αυτές τις περιοχές οι οποίες είναι υποένταξη τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο στον εκδημοκρατισμό, στο δικαστικό σύστημα, στην πάταξη της διαφθοράς και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σίγουρα διαπιστώνω από την έκθεση ότι υπάρχουν βελτιώσεις σημαντικές ε, σε όλα αυτά τα επίπεδα και όμως εξακολουθούν να υπάρχουν τα προβλήματα. Ε, τονίσατε το θέμα της ΦΥΡΟΜ και το θέμα της ε, Τουρκίας σε σχέση με τους γειτονές Και θα ήθελα να κάνω, για να μην καταχρώμε του χρόνου, να κάνω δύο ερωτήσεις ως προς αυτά. Βλέπετε σημεία υποχώρησης της κυβέρνησης της ΦΥΡΟΜ στο θέμα της συνεργασίας της με την Ελλάδα για την εξέβρεση λύσεως στο όνομα. Και ποια είναι αυτά. Δεύτερον, αν είπατε ότι υπάρχει μια βελτίωση των σχέσεων Άγκυρας Κύπρου Ποια είναι τα ορατά, διότι εγώ δεν έχω κάτι το ορατό, σημεία που δείχνουν ότι η Άγκυρα προσπαθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Πάκ για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, για κάθε χώρα εκθέσεις προόδου. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Και τα πέντε γενικά σημεία που μας υπενθυμίσατε. Είμαι ευγνώμων γιατί μερικοί τα έχουν ξεχάσει. Θυμίζω επίσης ότι και με ρώτησαν πριν μπω εδώ μέσα ότι δεν υπάρχει επίτροπος διεύρυνσης, πια τι θα γίνει ε, με εμά κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο αισιόδοξοι, να πούμε ότι η προκαταρρεκτική εργασία έγινε, κανείς δεν, σας, ε, ε, κανείς δεν θα σας την πάρει πίσω, ανεξάρτητα αν δεν υπάρχει επίτροπος διεύρυνσης, δεν χάνουν την προοπτική. Για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη πρέπει να πω ότι όλη η πολιτική στη Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι τόσο ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα του ποδοσφαίρου και αυτό Σημαντικό είναι ότι μέχρι τώρα ε, δεν μπορούσαν να ε, χαρούν όλοι για, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τα τελευταία δέκα χρόνια η συμφωνία του Ντέιτον χρησιμοποιεί το όλο και περισσότερο ε, για να αναδειχθεί αυτή η, η, η, η κρατική οντότητα και η ηθαγένεια. Ε, εγώ ε, είμαι, ε, χάρηκα με την κυρία Κορνέλησεν, η οποία σήμερα παραδέχτηκε ότι ψήφισε λάθος όταν ψηφίσαμε για την έκθεση. Τώρα χρειαζόμαστε κάποια κριτήρια και πώς θα γινόταν διαφορετικά ούτως ώστε να στους πολιτικούς εκεί. Εσείς κάνατε μία πρόταση για την αλλαγή μετά τις εκλογές έχασα το το εκλογικού, δικαίου, του, εκλογικού νόμου. Ε, αλλά τροποποιήθηκε ο εκλογικός νόμος ε, και Ε, συμφώνησαν πάρα πολύ. Μόνο ο Λαγκούμζα, ε, υπεύθυνο πολιτικός, δεν συμφώνησε. Πρέπει να του υπενθυμίσετε ότι ε, θα πρέπει να, για σε όλη τη Βοσνία Ερζεγοβίνη να δώσει μάχη για αυτούς που δέχονται την πρότασή του. Μιλήσατε λίγο περισσότερο γιατί έχετε διπλό όνομα ε, για το Φιρόμ τώρα. Ευχαριστώ και την αναφορά στη χώρα που έχω αναλάβει, ε, η οποία είπατε ότι παραμένει στο παιχνίδι, σε συνεργασία με το ε, κοινό ε, Βούλιο, ανανεώθηκε εντολή. Χάσαμε πολύ χρόνο με τη χώρα αυτή, η οποία τώρα ξαναγύρισε εκεί που ήταν τον περασμένο Δεκέμβρη και τώρα θα πρέπει να αναζωογονήσουμε τις ελπίδες τους χαιρετίζομαι την ένταξη της Κροατίας, θα πρέπει να εκτιμήσουμε και τον αντίκτυπο στα Σκόπια που είναι η χώρα με την μακρότερη ιστορία ε, καθεστώτος ε, χώρας ε, υποψήφιας που ακόμη περιμένει. Θα μπορούσε ο Επίτροπος να μας μιλήσει σχετικά με την πρόοδο με τα τις συστάσεις του συμφωνεί μαζί μου ότι η πολιτική βούληση χρειάζεται από όλες τις πλευρές και των εμπλεκομένων ε, στη χώρα αλλά χρειάζεται επίσης και συμβολή από τις γειτονικές χώρες. Επίσης ε, μπορούμε να χαιρετήσουμε την πρόσφατη δήλωση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικού ε, που ε, αναφέρεται στην, στο ενδεχόμενο μια συμφωνίας στα ενόψη και της ελληνικής προεδρίας. Θα πρέπει να υπάρξει έτσι νέα δυναμική για την επίλυση του προβλήματος του ονόματος. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει στις πρώιμες φάσεις των διαπραγματεύσεων, αν αρχίσουν τώρα, Νομίζω ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα του ονόματος. Επίσης η πρώτη εξέταση και το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 θα ε, κάλυπταν τις ανησυχίες των κρατών μελών για τη χώρα αυτή. Καλό είναι να εξετάσει το αίτημα αυτό ε, όταν θα συζητηθεί το θέμα και στις ε, πρωτεύουσες των κρατών μελών και των υποψηφίων κρατών. Και εσείς μακρηγορήσατε λίγο. Και τώρα ο κύριος Κασίν για τη Σερβία. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι βέβαιο πω η Κομισιόν και εσεί ε, προσωπικά, κύριε Επίτροπε, ε, κρατάτε μια δραστήρια στάση απέναντι στην ε, διαδικασία διεύρυνση. Πιστεύω πω αυτή η αξιολόγηση τη προόδου που έχουν σημειώσει το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η Ελβανία και το Κωσυφοπέδιο αντικατοπτρίζει την κατάσταση προόδου των χωρών, αλλά δίνει και μια ανεκτήμητη όθηση στι προσπάθειε των χωρών αυτών και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη που δεν εντάσσεται αυτό το πακέτο. Η αρχή τη εξομάλυση στο των σχέσεων ανάμεσα στη Σερβία και στο Κωσυφοπέδιο θα είναι πολύ δύσκολο να τη σκεφτεί κανεί χωρί την προοπτική τη ένταξη στην Ένωση. Ε, θεωρώ πως θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή τη ε, θετική φάση, χτυρώντας τη δική μας ε, πλευρά της συμφωνίας, ώστε να προχωρήσουν τα κράτη αυτά σε ένα υψηλότερο στάδιο ολοκλήρωση. Ε, επειδή είμαι εισηγητή για τη Σερβία, θα εστιάσω στα ε, επιτεύγματα τη κυβέρνηση του τελευταίου χρόνου. Αναμένω πω η αξιολόγηση της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου δεν θα αποκλίνουν για την πρόοδο της χώρας. Στην έκθεσή μου προς το Κοινοβούλιο τονίζω την ιστορική σημασία ε, συμφωνία των Βρυξελών ανάμεσα στην Σερβία και στο Κωσυφοπέδιο και είναι ήδη απόλυτα σαφές πως οι πολιτικοί ηγέτες των δύο χωρών αναγνώρισαν το διάλογο και την εξομάλυση των σχέσεων ως ε, συμφέρον και των δύο χωρών και θα συνεχίσουν σε αυτό το δρόμο. Στις, οι τοπικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στο Κοσφοπέδιο σηματοδότησαν ένα σημαντικό ε, ορόσημο. Ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις σημαντικές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν δύο χώρες, δηλαδή το κράτος δικαίου, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων. Ε, ε, θα ήθελα να καταδικάσουμε έντονα την ατυχή απόφαση για απογόρευση της παρέλασης ε, περηφάνειας στο Βελιγράδι. Θα πρέπει αντίθετα να εξασφαλίζει το, το κράτος δικαίου στη χώρα και η προστασία όλων των μειονοτήτων. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you. Κύριε ο Γιάννη για την Αλβανία. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Επίτροπο για την ε, εν γέννη θετική έκθεση περί διεύρυνσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την Αλβανία. Σας ευχαριστώ επίσης για τη διατύπωση που χρησιμοποιήσατε στην έκθεσή σας, στην εισήγησή σας, καθώς αυτή δείχνει την ε, προσήλωσή σας, την ε, αφοσίωσή σας στην επίδοση ανταμοιβή στις χώρες που κάνουν τις σωστές ενέργειες. Είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για την Αλβανία, που έχει κάνει τρομερές προσπάθειες και κινήσεις. Θυμάστε πριν από 20 χρόνια τους τραπεζίτες στην παραλία. Έχει, μια, έχει γίνει μια φυσιολογική ευρωπαϊκή χώρα. Εντάξει, μπορούν να γίνουν πράγματα για να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως έχουν γίνει βήματα μπροστά, βήματα προόδου και η στήριξη της Κομισιόν είναι πολύ σημαντική για όλα αυτά. Επίσης είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει και πάλι στον εαυτό της αλλά και στον κόσμο ότι είναι και θα είναι ένα στόχος, ότι υπάρχει κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε αυτή την Ήπειρο που θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το στόχο της. Πολύ συχνά στην Αλβανία ε, πολλές θεωρούμε ότι είναι πολύ άχρηστο όλα αυτά ή πολύ δαπανηρά. Αλλά τελικά φαίνεται πως αξίζουν τον κόπο. Όταν κανείς δει αντικειμενικά τα πράγματα, Η φετινή χρονιά ήταν πολύ καλή σε σχέση με τη διεύρυνση. Εγώ ως συζητητής είμαι ευγνώμων για την Κομισιόν για τις συστάσεις της και ειλικρινά ελπίζω πως θα εφαρμοστούν οι συστάσεις αυτές γιατί μιλάμε για εφαρμογή και ότι η Αλβανία θα μπορέσει να έχει καθεστώς υποψήφιας χώρας χωρίς άλλη καθυστέρηση. Φυσικά γνωρίζουμε πως οι απαιτήσει θα πρέπει να πληρώνται πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Όντως, ευχαριστώ. Η κυρία Όμαν, θα δώσω το καλό παράδειγμα συντομίας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ Επίτροπε. Είμαι ευγνώμων που δώσατε ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια της Κοπενχάγης. Θα ξεκινήσω επίσης με την εξή παρατήρηση. Είναι κρίμα που παρουσιάζεται σήμερα η έκθεσή σας, γιατί είναι Αγία Μέρα θρησκευτική μέρα σήμερα, είναι μάλλον αργία θρησκευτική στην Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τέλο πάντων, Επίτροπε, σα είπα και πέρυσι ότι η Τουρκία δείχνει δύο διαφορετικέ εικόνε και αυτό επιβεβαιώνεται και για το 2013. Από την θετική πλευρά είχαμε την μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματο, είχαμε τον πακέτο εκδημοκρατισμού της, της 30ης Σεπτεμβρίου όσον αφορά την γλώσσα και την ηθαγένεια. Έχουμε τις συνομιλίες με το ΠΚΚ, τον διαμεσολαβητή, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε ένα πολιτικό κλίμα όπου ο συμβιβασμός δεν φαίνεται να υπάρχει. Πολύ συχνά χρησιμοποιείται η προσέγγιση της απόλυτης ε, πλειοψηφίας και η πόλωση. Ο πρόεδρος Γκιούλ το μας προειδοποίησε γι' αυτό στις αρχές των εργασιών του Κοινοβουλίου. Έχουμε τις διαμαρτυρίες στην πλατεία Γέζη που τις καταδικάσαμε και εμείς την ε, αντίδραση ως Ευρωκοινοβούλιο. σε πραγματικές συνθήκες δημοκρατικές η πλειοψηφία πρέπει να λαμβάνει υπόψη την άποψη της μειονότητας και είναι ένα νόμο δικαίωμα ε, να μπορεί κανείς να διαμαρτυρηθεί. Και επίσης οι διαμαρτυρίες αυτές από την άλλη πλευρά μας έδειξαν ότι η Τουρκία ε, είναι μια ζωντανή κοινωνία που εκφράζει την άποψή της. Ωστόσο πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και την ελευθεροτυπία και τον πλουραλισμό που Τελευταία μου φράση. Όταν μιλάτε για ποδόσφαιρο, λυπόμαι που δεν τα κατάφεραν ε, χτες στις ε, κάτω χώρες ε, στο τελευταίο μάτς για το παγκόσμιο κύπελο αλλά να πω και ότι και τώρα πρέπει να παίξουμε μπάλα και στις σχέσεις με την Τουρκία η ευθυγράμμιση, ομαλοποίηση χρειάζεται. Mr. Rushek. Thank you, Chairman. Ο κύριος Ρούτσεκ. Επίτροπε, συνάδελφοι, νομίζω πως η πολιτική διεύρυνση είναι μια από τις πιο επιτυχίες πολιτικές που είχαμε που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο θα έλεγε πριν από 25 χρόνια ότι οι χώρε που ήταν πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα θα ήταν σήμερα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το λέω γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τι σημαίνει διεύρυνση. Ειρήνη, σταθερότητα, συνεργασία, ευημερία στις ε, περιοχές μας, στις περιφέρειές μας. Το 2013 ήταν επιτυχές έτος. Ε, ε, εντάχθηκε η Κροατία, διαπραγματεύεται το Μαυροβούνιο, υπάρχει πρόοδος στις σχέσεις ανάμεσα στο Βελιγράδι και την Πρίστινα, επιτυχής εκλογές και πρόοδος στην Αλβανία. Όσον αφορά το Σοσιαλιστική και Δημοκρατική Ομάδα, εμείς υποστηρίζουμε τη διαδικασία ε, διεύρυνσης στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε παρά τις δυσκολίες που έχουμε στα κράτη-μέλη μας. Θα συνεχίσουμε στην ίδια πορεία, γιατί δεν ξεχνάμε τι σημαίνει η διαδικασία διεύρυνσης. Ναι, οι χώρες και η πολιτική τους και οι δημόσιες διοικήσεις τους πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. υπάρχει μια πορεία για το τι πρέπει να κάνει κάθε χώρα. Και θα πρέπει να το κάνει. Και αυτό το υποστηρίζουμε. Αλλά επειδή είμαστε πολιτικοί, θα ήθελα επίσης να κάνω έκκληση σε εμά όλους. Και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Όταν δηλαδή μιλάμε για τη διεύρυνση, κάποιες φορές μιλάμε για τη διεύρυνση και στις χώρες μας. Και θα ήθελα να κάνω έκκληση σε εσά να συζητήσουμε τα θέματα με τους ανθρώπους μας, με το λαό μας, να χρησιμοποιήσουμε τις ευρωεκλογέ του χρόνου, ώστε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας τις χώρες μας και η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι τόσο ευνοϊκή και τόσο θετική προς τη διεύρυνση όπως και η σημερινή σύσταση. να πω ότι έχουμε μια ομάδα σοσιαλδημοκρατών από τις ε, ε, χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που καλέσαμε σήμερα για την ε, σημερινή περίσταση. Ήθελα να τους καλωσορίσω και βεβαίως να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Εξωτερικών που επέτρεψαν να είναι παρόντες σήμερα εδώ και να παρακολουθήσουν τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και μας ακούσατε. Ο κύριος Πρέντα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, για φέτος η Ισλανδία δεν έχει δικαίωμα μιας έκθεσης πρόοδου και όπως ξέρετε αυτή είναι η απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση μετά τις εκλογές του Απριλίου. Όπως ελέγχθη πολλές φορές, η Ισλανδία ήταν μια εξαιρετική υποψήφια χώρα και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προδικάσουμε τη συνέχεια. Ε, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει ε, ενδεχομένως θα ληφθεί μια απόφαση του Κοινοβουλίου ή θα γίνει λόγος για δημοψήφισμα. Εν πάση περιπτώσει, όπως ε, ελέγχ από τον Επίτροπο Φίλε και ε, με χαρά το, το λαμβάνουμε υπόψη. Η πόρτα παραμένει ανοιχτή για την Ισλανδία. Σας ευχαριστώ. Frau ε, Η κυρία Φλότρ, ευχαριστώ πολύ. Εγώ φοβάμαι ότι θα συμβεί το αντίθετο με αυτό που είπε ο κύριος Ρούτσεκ, γιατί νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μας εκστρατείας θα χρησιμοποιήσουμε το θέμα της ε, Τουρκίας, της υποψηφιότητας και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και βρίσκω ότι φέτος μας προτείνεται να ενεργοποιήσουμε πέρα από το κεφάλαιο 22 που αποτελεί το τέλος ενός ε, παγώματος των ε, διαδικασιών που διήρκησε μεγάλο χρονικό διάστημα να ξανανοίξουμε τα κεφάλαια 22 και 24 υποστηρίζοντας ε, α, που ελέγχθησαν σε σχέση με το πάρκο Γκεζί. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες είχαν δικαίωμα να διαδηλώνουν και να εκφράζουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερο μέσον από αυτό το μέσον της προσχώρησης που ε, επιτρέπει στις χώρες να προσχωρήσουν στο μέλλον. Πώς όμως να πείσουμε το Συμβούλιο για κάτι τέτοιο. Διότι σε επίπεδο Συμβουλίου θα πρέπει να μπορέσουμε να δράσουμε και να ανοίξουν τα κεφάλαια έτσι ώστε να ενισχύσουμε τη σχέση μας με την Τουρκία και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα στις σχέσεις μας, ε, στο θέμα της Συρίας, στο θέμα της ε, ε, ενέργειας γενικότερα και ας πω και στο δημογραφικό. Πώς θα πείσουμε το Συμβούλιο. Αυτό είναι το ερώτημά μου προς τον κύριο Φίλε. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε το κατάλογο των ομιλητών, να τελειώσουμε γιατί μας μένουν 8 ε, λεπτά και πρέπει να δώσουμε το λόγο να απαντήσει και ο Επίτροπος. Και αυτό είναι και το σωστό ερώτημα. Πώς θα, θα πείσουμε τα κράτη-μέλη να ε, γνωρίσουν, να συνειδητοποιήσουν την δυνατότητα που διανοίγεται. Ως προς την Τουρκία, θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής σε σχέση με ε, πέρσι, γιατί στην έκθεση πρόοδου το 12 σας είπα πώς είχαν τα πράγματα και η Επιτροπή είχε υπογραμμίσει την ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να προωθήσει τις ε, διαπραγματεύσεις για μια πλατφόρμα ε, προσχώρησης Τώρα βλέπουμε ότι η κυβερνητική οι Τούρκοι κυβερνητικοί και αξιωματούχοι μας βοηθούν σε αυτή την πορεία. Αυτό θα είναι και ένα από τα ε, θέματα που παραμένει ανοιχτό για το Συμβούλιο και ορισμένα κράτη-μέλη τονίζουν αυτές τις ε, δυνατότητες και ευκαιρίες που διανοίγονται. Μιλάμε για το άνοιγμα του κεφαλαίου 22. Αυτό δεν πρέπει να είναι μία ε, ad hoc όθηση στην διαδικασία προσχώρησης που θα περνάει η μία προεδρία στην άλλη. Έχουμε, έχουμε διανύσει τρία χρόνια και θα πρέπει να γίνει κάτι καλύτερο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ανοίξει το κεφάλαιο 22 να δούμε τις θετικές επιπτώσεις μιας θετικής ατζέντα και ελπίσουμε να έχουμε θετικά νέα ως προς τον ε, διάλογο θεωρήσεων και επανεισδοχής. Ανέφερα ότι η Τουρκία θα πρέπει να ανταποκριθεί στο συμπληρωματικό πρωτόκολλο. Μου μιλήσατε για κυρώσεις ε, η μεγαλύτερη κύρωση είναι ότι το Συμβούλιο έχει μπλοκάρει οκτώ κεφάλαια. Και σε αυτό συμφωνήσαμε ομόφωνα με βάση τις συστάσεις της Επιτροπής. Δεν είναι αυτή η πιο σοβαρή κύρωση. Όταν η Τουρκία ανταποκριθεί και συμμορφωθεί προς το συμπληρωματικό πρωτόκολλο θα ανοίξουν τα οκτώ αυτά κεφάλαια και αυτό θα αποτελέσει μια μεγάλη όθηση για τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα κεφάλαια 23 και 24 που θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο γιατί αν μιλάμε για τα γεγονότα του Μαΐου Ιουνίου που έλαβαν χώρα στην Τουρκία και θέλουμε να λάβουμε υπόψη ε, αυτό το αίτημα των πολιτών της Τουρκίας, ας χρησιμοποιήσουμε τα καλύτερα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, που είναι τα κεφάλαια 23 και 24. Σας υπενθυμίζω αυτά που ήδη ξέρετε. Δεν μπορέσαμε. Ούτε καν να ανταποκριθούμε στην ε, συγκριτική αξιολόγηση σε αυτό το benchmarking των ε, κεφαλαίων. Άρα θα δινόταν μεγάλη όθηση αν η ομάδα εργασίας για το κεφάλαιο 23 θα μπορούσε να ανοίξει τις διαπραγματεύσεις. Να ανοίξει δηλαδή αυτό το σημαντικό κεφάλαιο, το 23, ως προς την οριοθέτηση επιδόσεων. Ως προς ε, οριζόντια ζητήματα, ε, εκτιμώ την υποστήριξη των ε, εισηγητών και των συντονιστών. Θα ήθελα να σας εγγυηθώ το εξής. Η διαδικασία διεύρυνσης δεν βασίζεται σε έναν αυτόματο πιλότο, σε μία αυτόματη πλοήγηση. Βασίζεται σε εσά, με βάση μία διαδικασία ανάδρασης και αυτό που έχει σημασία είναι οι επιδόσεις και η αιρεσιμότητα. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο μπορούμε να προσδώσουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές καθαρά δεσμεύσεις των κρατών μελών. Γιατί έχει σημασία η διεύρυνση και δεν είναι ένα θέμα που αφορά τους επιτρόπους και τους βουλευτές, αλλά τους πολίτες των κρατών μελών. Γιατί με ενδιαφέρει η κοινή γνώμη ιδιαίτερα και ό,τι προσπαθώ να κάνω στη διαδικασία διεύρυνση τα τελευταία χρόνια με βάση αυτή την κινητήριο δύναμη είναι όχι να προβάλλω λέξεις αλλά και πολιτικές που να ενισχύσουν την αξιοπιστία της διαδικασίας διεύρυνσης. Όπως ξέρετε, με βάση την ε, τελευταία έκθεση προόδου για τη διεύρυνση το 2014 μιλούσαμε, το 2013 είχαμε αρχίσει να μιλάμε για αξιοπιστία, μετά μιλήσαμε για την διαδικασία μεταλλάξεων που ε, προβάλλεται μέσω των διαπραγματεύσεων διεύρυνσης. Τώρα μιλάμε για τα ουσιώδη, για τα θεμελιώδη ζητήματα και αυτό λέμε fundamentals first αυτό είναι το νέο μας σύνθημα. Μιλήσαμε λοιπόν για ζητήματα που αποτελούν τώρα αναπόσπαστο μέρος του κεκτημένου, αγνοώντας τις αλλαγές στις θέσεις ως προς την εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της οικονομικής διακυβέρνησης με βάση την προώθηση των ζητημάτων αυτών από τριμερείς διαλόγους και τις αντίστοιχες διαδικασίες διαθεσμικά. Γι' αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε αυτές τις πολιτικές, δηλαδή τα μακροοικονομικά ζητήματα, τα δημοσιονομικά ζητήματα. Μας ενδιαφέρει να υπάρχουν στοχοθετημένες πια συστάσεις και μια εποπτεία της εφαρμογής των συστάσεων. Πρόκειται για μια νέα πορεία που αφορά και την όλη διαδικασία συμμόρφωσης. Βλέπετε λοιπόν ότι βασιζόμαστε ε, στεναρά στο ε, θεσμικό πλαίσιο που προϋπάρχει και θα πρέπει μέσω αυτής της δημόσιας δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκριθούν οι χώρες αυτές για να μας δώσουν μία συνολική εικόνα των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που οδηγούν σε ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα έτσι ώστε οι υποψήφιες χώρες να αναλάβουν αυτή τη δράση και τις προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τις ίδιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τα κράτη-μέλη. Έτσι ώστε όταν προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι απόλυτα έτοιμες, όχι μόνο στα κεφάλαια 22, 23, 24, αλλά και σε όλους τους τομείς που αφορούν την οικονομική διακυβέρνηση. Ε, φύγει ε, το, βασικό αυτό ε, ερώτημα και εκφράστηκε ανησυχία από την Ιταλίδα βουλευτή για τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στη Μεσόγειο. Δεν θα ήθελα να πω να προβάλλω ένα επιχείρημα ότι α, εγώ ε, ασχολούμαι με την ε, διεύρυνση και με τίποτα άλλο. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Είναι ένα θέμα που αφορά ολόκληρο το Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ξέρετε ότι έγινε και πρόσφατα επίσκεψη στην ε, περιοχή αυτή. Δεν πρόκειται λοιπόν για ευθύνη ενός, δύο ή τριών κρατών. Πρόκειται για συλλογική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας διεύρυνσης οι χώρες που χτυπούν την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αναλαμβάνουν αυτή τη δέσμευση και τις υποχρεώσεις που έχουν έναντι ημών. Ως προς την Τουρκία και την Κύπρο. διαβλέπω νέα και θετικά στοιχεία, όχι μόνο σε επίπεδο λόγου και ρητορίας, αλλά έμπρακτα. Ο ειδικό εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών μίλησε για μια καινοτόμο προσέγγιση. Οι βασικοί, οι κύριοι διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές έχουν έχουν προσκληθεί στην Άγκυρα και στην Αθήνα και υπάρχουν περισσότερες, ε, ε, υπάρχουν, υπάρχει μεγαλύτερη διαδικασία ενθαρρύνσεων από τις αποφέ, επαφές που έγιναν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε έναν ειδικό εκπρόσωπο εκεί. Υπάρχει μία ε, ομάδα διαχείρισης στην Κύπρο και κατέστη σαφές υπό ποιου όρους θα μπορέσει να προωθηθεί το όλο ζήτημα και από αυτήν την steering group. Ως προς την Βοσνία Ερζεγοβίνη και την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έχει συσταθεί μία ομάδα η οποία προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει τις θετικές συζητήσεις που έγιναν την 1η και 10η Οκτωβρίου μέσα στα πλαίσια του Γενικού Διαλόγου της ε, διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την ε, μελλοντική προσχώρηση. Ελπίζω να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις χώρες να φτάσουν σε μια συμφωνία έτσι ώστε να αλλάξει το σύνταγμα της χώρας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην ετοιμιγορία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής διαδικασίας και μεταρρυθμίσεων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές όμως ότι αυτό δεν θα γίνει εις βάρος της ετοιμιγορίας του ΕΔΑΔ οι επικεφαλείς, οι ηγέτες της Βοσνίας εσρεγοβίνης θα πρέπει να κατανοήσουν ότι θα πρέπει να διανύσουν αυτή την απόσταση μεταξύ των συμφωνιών του Dayton και της ε, διεύρυνσης. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σωρία ζητημάτων και δεν αναφέρθηκα σε όλα θα πρέπει να μπορούν να ομιλούν με μία ε, φωνή για, σε επιμέρους ζητήματα. Και θα έπρεπε να βοηθήσουν τη διαδικασία ε, της προσχώρησης και της Κροατίας, να υποβοηθήσουν αυτή τη διαδικασία μέσω του προενταξιακού μέσου. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η γεφύρωση του χάσματος έτσι ώστε να περάσουμε από το Dayton, από τη συμφωνία του Dayton στην ε, προενταξιακή διαδικασία. Υπάρχουν ε, πολλές ε, συνέπειες βεβαίως αν κανείς δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις του και αυτό το τόνισα και μίλησα και για τις διαδικασίες μέσα στα πλαίσια του προενταξιακού μέσου για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη για να μπορέσει να ανταποκριθεί και σε άλλες ανάγκες της περιοχής. Ελπίζω να ανταποκριθούν και από πλευράς κινήτρων που δίνουμε και από πλευράς καρότου δηλαδή έτσι ώστε να να μπορέσουμε να, τους, να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα περισσότερο και στα επιμέρους ζητήματα της διαδικασίας αυτής. Ως προς την πρώην δημοκρατική, ε, ως προς την ΦΥΡΟΜ, πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, χάσαμε πολύ χρόνο. Και με ανησυχεί η νέα έκθεση ως προς την τύχη της ομάδας εργασίας για τις συστάσεις ε, της Επιτροπής. Ποια είναι η έκφαση δηλαδή του όλου ζητήματος. Και ελπίζω και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να προωθήσουν αυτό τον διάλογο που δεν θα θέσει ένα αμφιβόλο αυτή τη συμφωνία και την εφαρμογή της. Και ελπίζω η κυβέρνηση και πάλι να ξαναδεί τους όρους σε σχέση με το θέμα των σκοπίων, της κατάστασης των σκοπίων. Όταν μιλάμε για την εκλογική διαδικασία δηλαδή της ε, ε, φύρων, να μπορέσουν δηλαδή τα σκόπια να ανταποκριθούν σε αυτή τη ε, διαδικασία Έχουμε λάβει υπόψη τα ευρήματα της Επιτροπής αυτής της ομάδας αυτής ως προς την έκθεση προόδου και ελπίζουμε η κυβέρνηση να είναι σε θέση, στη θέση να προωθήσει έναν επικοδομητικό ε, διάλογο και με την Ένωση Δημοσιογράφων. Με βάση τη Συμφωνία της 1ης Μαρτίου, και ελπίζω η Ένωση Δημοσιογράφων και Συντακτών να κάνει τη βέλτιστη δυνατή χρήση αυτού του διαλόγου και να λάβει επικοδομητική στάση προωθώντας αυτό το διάλογο με τις αρμόδιες αρχές. Συμφωνώ με εκείνους που ανέφεραν ότι η ελληνική προεδρία είναι, αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για ολόκληρη την ε, περιφέρεια και προς τις ελληνικές αρχές έκανα μια προτροπή ιδιαίτερα προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πείτε μας πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας να βοηθηθούν όλες οι χώρες της ευρύτερης περιφέρειας και όχι μόνο μερικές. Δηλαδή να προχωρήσουν προς την ευρωπαϊκή τους ενταξιακή φιλοδοξία. Και αυτό ακριβώς προτείναμε και φέτος στη Φύρομ. προωθώντας το ζήτημα προς όλες τις χώρες να υπάρξουν εγγυήσει και χέγγια ότι η περσινή πρόταση είναι μια βιώσιμη πρόταση η οποία θα οδηγήσει σε καλύτερους όρους για να ασχοληθούμε και με το ζήτημα της ονομασίας και να το αντιμετωπίσουμε θετικά. και το μήνυμα προς τους πολιτικούς αφορά και ζητήματα χρονισμού και όχι αντιτίμου σε ένα συμβιβασμό. Αλλά να δούμε αυτό το status quo αποδίδει, ποιο είναι το τίμημα αυτού του status κουβό. Να μην χρονοτριβούμε δηλαδή, γιατί υπάρχει πάντα ένα εμπλεκόμενο κόστος σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως δεν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Προσπάθησα όμως, πολύ καλές και εύστοχες ήταν όλες οι ερωτήσεις και είπε και ο πρόεδρος ότι μετά την ε, παρουσίαση αυτή θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να επανέλθουμε σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα, αλλά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την υποστήριξη της Επιτροπής σας και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους οποίους συνδιαλέγομαι κάθε μέρα. Ευχαριστώ. Session is closed. συνεδρίασης. Thank